Εγώ ψήφισα και τράβηξα ίσως πολύ γρήγορα την κάρτα μου. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχει καταγραφεί η ψήφος μας. Θα το ελέγξουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, από το ε, ΕΛΚ και από το, τους σοσιαλιστές έχω λάβει τις εξής παρακλήσεις να τοποθετηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο κύριος Σούλμας, μεταφορών Άνταμ Κόσα και ε, Γεωργία Ερή Καντριό. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, επιβεβαιώνονται αυτές οι αλλαγές το πρακτικά θα